Ε, να τοποθετηθεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ο κύριος Σούλμας, Μεταφορών Άνταμ Κόσα και ε, Γεωργία Σερίκ Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ε, επιβεβαιώνονται αυτές οι αλλαγές. Το πρακτικά θα υιοθετηθούν στην επόμενη συνεδρίαση και ε, ε, ε, συμφωνείτε θα ειδοποιήσω τους συντάκτες των ψηφισμάτων για το αποτέλεσμα. Διακόπτεται η συνεδρίαση. Σας εύχομαι σε όλους